Δεκέμβριο του 2010 ως παγκόσμιο μερίδιο, ενώ ταυτόχρονα το δολάριο των Ηνωμένων Πολιτειών και το γεν έχουν μειώσει τα μερίδια τους σημαντικά σε ό,τι αφορά στα συναλλαγματικά αποθέματα. Αντίστοιχα μπορεί κανείς να διαπιστώσει και ως προς τη συναλλακτική αξία του ευρώ ή την ε, αξία ε, στην οποία εκδίδονται ε, ομόλογα. Είναι λοιπόν ε, επιτυχής ιστορία του ευρώ. Από την άλλη έχουμε όμως κρίση χρέους ορισμένα κράτη της Ευρωζώνης που συνδέονται με ευάλωτο ε, χρηματοοικονομικό τομέα και έλλειψη ανταγωνιστικότητας σε ορισμένες χώρες. Αυτή η κρίση τόνισε μια σειρά προκλήσεων που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο ιστορικό της Ευρωζώνης. Ορισμένες είναι βραχυπρόθεσμες, άλλες μέσοπρόθεσμες. Πρόκληση παριθμών 1. Πώς θα αντιμετωπίσουμε την ε, πιθανή αρνητική επίπτωση ε, μεταξύ ε, Τη ε, κρίση ε, του δημόσιου χρέους, του χρηματοπιστωτικού τομέα και τη πραγματικής οικονομίας. Είναι ένα τρίγωνο. Το βασικό ερώτημα είναι η σχέση όμως μεταξύ νομισματικής πολιτικής και χρηματοοικονομικής σταθερότητα. Υπάρχει μια σαφή ιεράρχηση στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με αυτού του στόχου. Ταυτόχρονα αυτό όμω δεν σημαίνει απαραίτητο ότι ε, θα πρέπει το ένα να υποκαταστήσει το άλλο. Ε, χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να καταλάβουμε καλύτερα το ρόλο που διαδραματίζει ο χρηματοοικονομικός τομέας στο ε, νομισματικό μηχανισμό. Είναι πολύ σημαντικό να ε, το καταλάβουμε. Οι φούσκες των τιμών στην αγορά και στη χρήματα χρηματαγορά τονώθηκαν και φούσκωσαν πραγματικά για πολύ καιρό και αυτό δεν το είχαμε αντιληφθεί ως πρόβλημα νομισματικής πολιτικής για μεγάλο διάστημα. Πρόκληση παριθμών 2. Η κρίση κατέδειξε σαφέστατα ότι η οικονομική διακυβέρνηση στην ΟΝΕ είναι και παραμένει πολύ ασθενής. Ή να το πω γενικότερα. Το σημερινό καθεστώς της Νομισματικής Ένωσης, χωρίς δημοσιονομική και πολιτική ένωση, ε, συνιστά ένα εύθραυστο κατασκεύασμα. Ε, πρόσφατα εγκρίθηκε η δέσμη των έξι νομοθετικών ε, ε, προτάσεων για να ενισχυθεί ε, το Σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη. Χρειάζεται όμω να ακολουθήσουν και άλλα βήματα για να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα τη ευρωζώνη στο σύνολό τη. Η εντολή τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα πληγεί αν ακολουθήσουμε αυτή την ατραπό. Ωστόσο, άλλοι ενεχόμενοι ε, θα επηρεαστούν περισσότερο. Το θέμα που διακυβεύεται εδώ λοιπόν είναι περισσότερο δημοσιονομική, άρα και πολιτική ολοκλήρωση. Πρόκληση υπαριθμών 3 το ζήτημα τώρα είναι και το ερώτημα πότε και πώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να επαναπροσαρμόσει τη νομισματική της πολιτική και να σταματήσει τα έκτακτα μέτρα που έλαβε για να ανταποκριθεί στην κατάσταση και να επανέλθει σε μία ομαλότητα. Αυτό αφορά το SMP που είναι ε, ένα σύστημα προσωρινό, περιορισμένο και αποστηρωμένο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρόσφατα φάνηκε και αναδύθηκε ως ο μόνος ε, φορέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη που μπορούσε να δράσει γρήγορα και αποφασιστικά. Το θέμα λοιπόν είναι τι πρέπει να γίνει στην υπόλοιπη Ευρωζώνη έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μην είναι το μόνο θεσμικό όργανο σε θέση να δράσει τέτοιες περιστάσεις. Και τι πρέπει να συμβεί έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σιγά σιγά ε, και μάλιστα το συντομότερο ε, να ε, καταργήσει τα έκτακτα μέτρα και να επιστρέψει στην ομαλότητα μόλις το επιτρέψουν οι αγορές. Η σειρά που πρέπει να γίνει αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμη, ιδιαίτερα στο παρόν οικονομικό περιβάλλον που έχουμε όλο και περισσότερους κινδύνους. Αντιμετωπίζοντας λοιπόν όλες αυτές τις προκλήσεις, θα έλεγα ότι οφείλουμε να λάβουμε υπόψη μας ότι η Ευρώπη δεν είναι νησί. Κανείς δεν είναι νησί σε αυτόν τον κόσμο. Ακόμα και αν η παρούσα κρίση μας έχει κάνει πάρα πολύ εσωστρεφείς. Θα πρέπει να ε, τοποθετηθούμε παγκοσμίω σε συνεργασία με τους ε, γείτονές μας, αλλά και σε ανταγωνισμό με άλλες μεγάλες ανεπτυγμένες ή αναδυόμενες οικονομίες. Αυτό έχει να κάνει με όλους τους τομείς πολιτικής, με και της νομισματικής πολιτικής. Η συνεργασία θα πρέπει να αυξηθεί σεβόμενοι πάντα διαφορετικές αφετηρίες, διαφορετικές εντολές και διαφορετικό ιστορικό υπόβαθρο. Όλοι υπό αυτή την έννοια έχουμε κοινέ μεν πλην διαφορετικές ευθύνες. Δεδομένης της εκπαίδευση και επαγγελματική μου κατάρτισης θεωρώ ότι έχω τα προσόντα και τα εφόδια για να συνεισφέρω να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις που σας περιέγραψα μόλις. Ε, στα διοδρομία μου επαγγελματικά ε, είχε εστιαστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωζώνη και τη διεθνή οικονομική διακυβέρνηση από διάφορε σκοπιές έκανα ε, μεταπτυχιακό στην οικονομία μάστερ στο Πανεπιστήμιο της ΒΟΝ στη Γερμανία σε θέματα νομισματικά και συναγματικών ε, ισοτιμιών, MBA στο Πανεπιστήμιο Βοκόνη στην Ιταλία και ε, άρχισα τη σταδιοδρομία μου σε μια ιδιωτική συμβουλευτική εταιρεία στην Κολονία, όπου μεταξύ άλλων συμμετείχα σε προγράμματα ΦΑΡ στην Ουγγαρία, στις χώρες της Βαλτικής και στην τότε ακόμα Τσεχοσλοβακία. Το 1996 άρχισα να εργάζομαι στο Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών, όπου και μέχρι σήμερα βρίσκομαι. Η πρώτη μου θέση ήταν στο τμήμα Παγκόσμια Οικονομία, Νομισματικά Θέματα και G-Groups, που τότε G ήταν κυρίως η G7. Ε, ε, είχα ασχοληθεί με ασιατικές χώρες, ιδιαίτερα την περίοδο της ε, ασιατικής κρίσης και στη συνέχεια προσωπικός βοηθός του Γενικού Γραμματέα και ε, αργότερα ε, επικεφαλής του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Υπουργού. Έχω ασχοληθεί με θέματα ευρωπαϊκά. Το Μάρτιο του 2003 ανέλαβα ως Γενικός Διευθυντής ε, στο τμήμα Χρήματα Αγορών που τότε συμπεριλάμβανε και διεθνή ζητήματα. Η εποπτεία αφορούσε την KFW Banking Group, το γερμανικό οργανισμό αντιμετώπισης κρίσης και την BaFin. G7, G8, G20, όλα αυτά ήταν θέματα που έχω χειριστεί το Διεθνές Δομισματικό Ταμείο και οι σχέσεις μας με χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2008 ανέλαβα υφυπουργό ε, αρμόδιος για θέματα οικονομικά χρήματα αγορών. Είμαι μέλος σε διάφορες επιτροπέ υψηλού επίπεδου και για τους G20, G7, UFC, Euro Working Group, το Διοικητικό Συμβούλιο του EFSF και ε, του χρηματοπιστωτικού ε, συστήματος σταθερότητας. Επίσης, εκπρόσωπος ε, της Γερμανίας ε, στην Παγκόσμια Τράπεζα και την Τράπεζα Νοικοδόμησης και Ανάπτυξης. Είμαι μέλος ε, του Διοικητικού Συμβουλίου της Deutsche Telekom και της Γερμανικής Υπηρεσίας για Τεχνική Συνεργασία στην Αναπτυξιακή Βοήθεια. Επίσης προείσταμε στο Εποπτικό Συμβούλιο της εταιρείας Buffin και σε μια άλλη δομή για τη σταθεροποίηση των αγορών. Το 2011 ε, ήμουν ο ΣΕΡΠΑ της ε, κυρίας Μέρκελ στο G20 και μαζί με τον Μεξικανό συνάδελφο ε, συμπροέδρευσα στην ομάδα εργασίας του G20 για την μεταρρύθμιση του διεθνούς χρηματοπιστωτικού, νομισματικού μάλλον συστήματος. Μετά την κατάρρευση της τράπεζας Lehman Brothers το 2008 μαζί με τον Γένς Βάιτμαν και τον Άξελ Βέβερ ε, συντόνισα την απάντηση της γερμανικής κυβέρνησης στην κρίση, σταθεροποίηση της τράπεζας, Hippo Real Estate. Ε, σχεδιάσαμε το νόμο για τη σταθεροποίηση των αγορών και ιδρύσαμε τον αντίστοιχο οργανισμό. Από τότε που ξέσπασε η κρίση χρέους, συμμετείχα πάρα πολύ έντονα στην αντιμετώπιση της κρίσης και στη διαχείριση και στην ίδρυση του EFSF και στην αντιμετώπιση ε, της Ευρωζώνης και το Συμβούλιο και ορισμένοι θα θεωρούν φυσιολογικό όταν κάποιο περιαυτολογεί τόσο πολύ και αναφέρεται συνεχώ στον εαυτό του, είναι αρνητικό. Γνωρίζω ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν γίνει με μια ομάδα με πολύ μεγάλη προσήλωση και αφοσίωση. Δεν θα μπορούσαν να είχαν γίνει όλα αυτά χωρί αυτή την ομάδα των συνεργατών που με πλαισιών. Δεν τα έκαναν μόνο, μόνος μου. Πάρα πολλοί ε, ήταν εκείνοι που με βοήθησαν και με στήριξαν σε αυτή την προσπάθεια. Ολοκληρώνεται, λέει η Πρόεδρος, μάλιστα. Σύντομα, θα ήθελα να αφαιρθώ στα εξή δύο, αν μου επιτρέπετε. Μπορεί να πείτε ορισμένοι ότι εγώ δεν έχω εμπειρία σε κεντρική τράπεζα. Προφανώς. Ισχύει αυτό. Αλλά καθ' όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου ήμουν σε στενή επαφή με την Κεντρική Τράπεζα και τον αντίστοιχο κόσμο, γιατί στη Γερμανία ε, είναι κοινή η ε, ευθύνη και για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και για την εποπτεία των τραπεζών και το θέμα του G20 και G7 είναι μια κοινή ομάδα ε, όπου συμμετέχουν οι εκπρόσωποι και του Υπουργείου Οικονομικών και της Κεντρικής Τράπεζας και από την ε, ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας συνεργάζομαι με το προσωπικό της. Γνωρίζω λοιπόν τον πολιτισμό και την κουλτούρα μιας Κεντρικής Τράπεζας αρκετά για να εργαστώ εκεί. Αλλά επίσης πιστεύω ότι μπορεί να είναι προστιθέμενη αξία στο ε, Διοικητικό Συμβούλιο η πρώτερη εμπειρία σε κάποιο διαφορετικό κλάδο. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για μένα είναι η επικοινωνία. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να ανακοινώνει τη στρατηγική τη τι αποφάσει τη στους Ευρωπαίους πολίτες και στου εκπροσώπου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και πιστεύω ότι πραγματικά αυτό είναι κομβικό για να διατηρηθεί το σημαντικότερο, το πιο πολύτιμο αγαθό που έχει κάθε κεντρική τράπεζα και είναι η αξιοπιστία αυτή. Ο στόχος της επικοινωνίας είναι βεβαίως ε, περίπλοκη υπόθεση μια μοναδική ενιαία νομισματική πολιτική αντιμετωπίζει τους πολίτες στα 17 κράτη-μέλη με διαφορετικό πολιτικό και οικονομικό υπόβαθρο και πραγματικότητα και διαφορετική ιστορία, γλώσσα και κουλτούρα κάθε φορά. Ταυτόχρονα η σημασία του ενιαίου νομίσματος σημαίνει ότι οι παγκόσμιες χρηματαγορές ακούνε προσεκτικά αφού κράζονται. Αυτός ο συνδυασμός καθιστά απόλυτη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μιλεί με μία φωνή. Συμπεραίνοντας, θα ήθελα να πω ότι αντλούοντας από την εμπειρία μου και τις γνώσεις μου ε, θέλω να συνεισφέρω ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τη ΕΚΤ στην ευημερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα της Ευρωζώνης και των πολιτών της με μία εντολή και εντός τη εντολή που έχει δοθεί στην ΕΚΤ, δηλαδή κατά κύριο λόγο η διατήρηση τη σταθερότητα των τιμών. Επιθυμώ όλα αυτά να τα προσφέρω με σαφή προσήλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη συνολικά ως κάποιος που είναι κάτοχος γερμανικού διαβατηρίου αλλά γνωρίζοντας την οικονομική και πολιτική κατάσταση στην Ευρώπη και με ε, ακλόνητη πρόθεση να υπηρετήσω τον Ευρωπαίο πολίτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάμε στον επόμενο γύρο ερωτήσεων. Πρώτα εκ μέρους του ΕΛΚ, Βέρνα Λάγκεν. Ναι, όχι. Ο Ζαν Πολ ξανά. Καλώς δεν άλλαξε ο κατάλογος. Λοιπόν, ο Ζαν Πολ έχει το λόγο. Ζητώ συγγνώμη για το μπέρδεμα. Όχι, δεν άλλαξε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε μου σε αυτή την Επίτροπη για να δεχτείτε τα πειρά των ερωτήσεων. Ε, είπατε κάποια πράγματα στην παρουσίασή σας που μου ήταν ευχάριστα και κυρίως ότι δεν υπήρχε πραγματική κρίση του ευρώ σήμερα είναι κάτι που θα πρέπει στην προσπάθεια επικοινωνίας που θέλετε να κάνετε να επαναλαμβάνετε. Να σας θέσω ένα επίκαιρο ερώτημα. Χθε η Γερμανίδα Καγκελάριος και ο Γάλλος Πρόεδρος συναντήθηκαν για μία ώρα και μετά σε δείπνο μίλησαν για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ε, είπαν ότι συμφωνούν επί της αρχής αυτής της ανακεφαλαιοποίησης αλλά οι λεπτομέρειες δεν δόθηκαν, θα χορηγηθούν σε κάποιο χρονικό διάστημα. Έχω δει ερώτηση. Πρώτα απ' όλα, τι σκέφτεσαι για την ανάγκη, μία ανάγκη κεφαλαιοποίησης των Ευρωπαϊκών Τραπεζών. Δεύτερον, ε, πιο δισταμένο θέλετε, πιστεύετε ότι είναι καλή μέθοδος να ανακοινώνονται αρχές που δεν εφαρμόζονται άμεσα ούτως ώστε οι αγορές ίσως για μία ακόμη φορά να διαταράσσονται. Ευχαριστώ. Απάντηση. Καταρχάς, εν συντομία, να πω ότι δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Θα πρέπει να το λέμε πιο επανειλημμένα και πιο δυνατά ότι δεν έχουμε κρίση του ευρώ, δεν αληθεύει και δεν υποστηρίζεται από αποδείξει γεγονότα. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερα. Πρέπει να πούμε περηφάνεια ότι έχουμε ένα ισχυρό και σταθερό νόμισμα και να το λέμε σε όλο τον κόσμο αυτό. Αναφερθήκατε σε μια συνάντηση του Γάλλου Προέδρου και της Γερμανίδας Καγκελαρίου που έλαβε χώρα χθες. Ναι, είναι καλή αφετηρία αυτή να υπάρξει η γαλλογερμανική συμφωνία. Είναι κάτι αναγκαίο, είναι αναγκαία, όχι όμως επαρκής προϋπόθεσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν καλό αυτό που έγινε χθε. καλή αφετηρία, αλλά θα πρέπει να απευθυνθεί προς γείτονες και προς εταίρους κάποιος. Αναφερθήκατε στην επανακεφαλοποίηση των τραπεζών και είπατε κάποιες λεπτομέρειες. Θα έλεγα ότι θα πρέπει αυτό να είναι ένα στοιχείο από ένα πλήρες πακέτο το οποίο θα πρέπει να ετοιμάσουμε για την Ευρωζώνη και κυρίως για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση στην Ελλάδα ένα στοιχείο που δεν θα πρέπει να θεωρηθεί απομονωμένα. Κανένα απομονωμένο εργαλείο δεν θα μας βοηθήσει. Θα πρέπει να αποφασίσουμε για ένα πακέτο να αποφασίσουμε πρώτα απ' όλα και μετά να γίνουν λειτουργικά αυτά τα μέσα με τη σωστή σειρά. Ένα συνολικό πακέτο λοιπόν χρειάζεται που θα πρέπει να συνδυάζει πέντε στοιχεία. Πρώτα απ' όλα μια αξιόπιστη λύση για την Ελλάδα. Δεύτερον, αν χρειαστεί να δημιουργήσουμε κάποια τύχη προστασίας, δηλαδή να ενισχύσουμε το μέσο ε, ε, ενίσχυσης το EFSF για να περιοριστεί η διάδοση του φαινομένου και να κάνουμε αποτελεσματικότερη χρήση της δυνάμεως πυρός του EFSF. Τρίτον, ναι, και άλλο ένα μέσο είδη τείχους είναι η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση των τραπεζών σε χρηματοδότηση, κυρίως βράχη πρόθεσμη χρηματοδότηση. Αυτό θα πρέπει να γίνει σε ένα πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ενώση των 27 κρατών μελών για να αποφύγουμε στιγματισμό κάποιων καλύτερα να μην γίνεται από κάθε θεσμικό όργανο ξεχωριστά αλλά για όλες τις θυμικά σημαντικές τράπεζες των 27 κρατών μελών να γίνει αυτό ταυτόχρονα. Τέταρτον, του συνολικού πακέτου, τέταρτο σημείο του συνολικού πακέτου, δέσμευση για πιο ορθή οικονομική και φορολογική πολιτική που θα ακολουθείτε στις χώρες αυτές, τις χώρες που έχουν πρόβλημα και αυτές που ενδεχόμενο να πληγούν πια στο φαινομένο και τρίτο πιο μακροπρόθεσμα να υπάρχει καλύτερη διακυβέρνηση ε, της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης πιο μακροπρόθεσμα που θα απαιτεί και αλλαγή των συνθήκων. Άρα για να απαντήσω στο ερώτημά σας, είμαι υπέρ ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών αυτό σαν ένα κομμάτι ευρύτερου γενικότερου πακέτου, όχι σαν κάτι που είναι μεμονωμένο, σαν μεμονωμένο εργαλείο. Αν με ρωτάτε αν είναι καλή στρατηγική που χτες έγινε συνέντευξη τύπου Χρειάζεται χρόνο είναι η απάντηση για την επεξεργασία αυτών των γενικών πακέτων. Η Γενική Συμφωνία ήταν κάτι επικοδομητικό, αυτό που έγινε χτε. Τώρα χρειάζεται επεξεργασία λεπτομέρειε. Μέχρι τη διεξαγωγή τη Συνόδου Κορυφή στι 23 Οκτωβρίου. Thank you very much. Uh, next on behalf... Επόμενη, νομίζω, Αντελίν είναι ο επόμενος, εκτός αν έχετε αλλάξει τη σειρά. Ο Αντολίν Σάντσες Πρεσέδο. Okay, so you, you, you are going first. Πρώτο ο Μπούλμαν. Sharon, you are mixed up when it comes to the big groups in the house. I know that. Ξέρω ότι όταν γίνεται Λόγο για τι μεγάλε πολιτικέ ομάδε, καμιά φορά προκαλείται σύγχυση. Μην ενισχύετε. Λοιπόν, κύριε Άσμουσεν, σα καλωσορίζουμε εκ μέρου τη Σοσιαλδημοκρατική πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θέλω να αναφερθώ σε ένα θέμα το οποίο ε, στι γραπτέ απαντήσει που δίνεται αναφέρεται επανειλημμένα. Πρόκειται για το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Δηλαδή τόσο στο βιογραφικό σα όσο και στη δουλειά που κάνετε τώρα αλλά και στο πολιτικό σα όραμα παραπέμπεται του στην ομάδα των G20 πολύ καλά ακούγεται αυτό. Θέλω όμω ε, να γνωρίζω τι ακριβώ εννοείται. Ε, σε τι επίπεδο παραπέμπεται. Μιλάμε για την νομισματική πολιτική. Ε, θυμάμαι πριν από την κρίση ο κύριο Μπόφιγκα οποτεδήποτε έλεγε ότι οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες πρέπει να παρεμβαίνουν για να στηρίζουν τα νομίσματα, αυτό εννοείται ή μήπως μιλάτε για ρυθμίσεις, ρυθμίσεις και εποπτεία ε, μετά την κρίση οι G20 πολλοί λένε ότι θα πρέπει να αναλάβουν μια τελείως διαφορετική θέση. Τώρα λοιπόν ε, που πρόκειται να φύγετε από τη Γερμανία μήπως ε, θα μπορούσατε να είστε και κάποια φορά φιλοξενούμενος δικός μας οποτεδήποτε συζητάμε με το Συμβούλιο για τον έλεγχο των hedge funds ή οτιδήποτε άλλο. Φαντάζομαι ότι και με τη νέα ιδιότητα που θα έχετε θα έχετε χρόνο να είστε φιλοξενούμενος αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ θέλω να, ε, να επισημάνω το εξή. κάτω το παρελθόν ε, τα κράτη-μέλη δεν το ήθελαν αυτό. Είχαν μπλοκάρει το να μπορεί η ομάδα των G20 να παίζει αυτό το ρυθμιστικό ρόλο. Πώς μπορούμε λοιπόν να το αλλάξουμε αυτό. Πώς μπορούμε να βρούμε μια λύση για ένα κράτος μέλος, αναφέρουμε στην Ελλάδα, που δεν έχει ούτε το ίμιση του προϋπολογισμού της Βαβαρίας. Και ε, δεν έχουμε πείσει κανέναν μέχρι τώρα. Γιατί λοιπόν πιστεύετε ότι το Μάτων G20 θα μπορούσαμε ενδεχομένω να του εντυπωσιάσουμε. Απάντηση. Ε, φαντάζομαι να μην σας ενοχλεί που θα απαντήσω στα αγγλικά ε, και ελπίζω να έχουμε στο μέλλον περισσότερες ευκαιρίες να ε, συναντηθούμε εξαρτάται από το αποτέλεσμα της σημερινή ημέρα, το τι θα προκύψει μετά την ακρόασή μου. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι όσον αφορά αυτή τη διαδικασία των G20 εγώ της αποδίδω ιδιαίτερη σημασία. Ξέρετε γιατί, γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Ξεκίνησε το 99 στο Βερολίνο σε επίπεδο κεντρικών ε, τραπεζών τραπεζιτών και υπουργών οικονομικών και μετά ανοίχθη σε ανώτερο επίπεδο, αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων λόγω της κρίσης. Το G20 λοιπόν είναι το ανώτατο φόρουμ οικονομικής διακυβέρνησης και απέδειξε ότι είναι ένα πολύ αποτελεσματικό φόρουμ κυρίως σε περιόδους κρίσης και όπως πολύ σωστά υπενηχθήκατε τώρα η ομάδα G20 πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να αποδώσει, ότι μπορεί να ορίσει ένα παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό πλαίσιο που θα είναι εποφελές για τους πολίτες, για τους πολίτες των κρατών και της Τουντζίκος και περαιτέρω. Υπάρχει λοιπόν μία συζήτηση κατά πόσον ε, οι 20 είναι ο σωστό αριθμό, ε, κατά πόσον οι χώρες που λαμβάνουν σε αυτήν την ομάδα είναι οι σωστές χώρες. Εμείς δεν βλέπουμε να υπάρχει καμία διάσταση ανάμεσα στην νομιμότητα και την αποτελεσματικότητα που χαρακτηρίζουν αυτήν την ομάδα. Μάλλον, να το πω αλλιώ, είναι αποτελεσματική, αλλά ίσω πια να μην νομιμοποιούνται απόλυτα λόγω του ότι έχει αλλάξει και η δομή τη αγορά. Θα πρέπει να είναι περισσότερα τα κράτη που θα ε, συμμετέχουν στη χώρα αυτή και αυτό θα τους καθιστά και κατά 100% νόμιμους και 100% αποτελεσματικούς. Όσον αφορά την ομάδα G20 υπάρχουν δύο τομείς. Υπάρχουν τα νομισματικά ε, και υπάρχουν και τα χρηματοψηφιακά, τα δημοσιονομικά. Ε, υπάρχουν και άλλα θέματα που αφορούν την ομάδα των G20. Δεν πρέπει όμως να επεκτείνουμε αυτή τη βεντάλια, να την ανοίξουμε τόσο γρήγορα. Πρέπει καταρχήν να είμαστε αποτελεσματικοί σε αυτά που υποσχοθήκαμε. Όσον αφορά τώρα τα θέματα που χρήζουν ρυθμίσεων ε, σε χρηματοπιστωτικό επίπεδο. Νομίζω ότι έχουν γίνει πάρα πολλά, κυρίως μετά τη συνάντηση κορυφή στο Πίτσμπουργκ, αλλά χρειάζεται μεγάλο χρονικό διάστημα Νομίζω σήμερα το απόγευμα αργότερα θα έχετε τον τρίλογο για την έννοια. Μέχρι το 2012 ε, στο Πιτσμπουργκ ε, ανελήφθη μία υπόσχεση ε, ότι θα προχωρήσει το θέμα. Υπάρχουν πολύ προχωρημένες νομοθετικές προτάσεις σε χώρες Ασίας. Δεν έγιναν και πάρα πολλά πράγματα, ούτε και στη Λατινική Αμερική. Κατά κάποιον τρόπο λοιπόν έχουμε χάσει το δυναμισμό μας ε, σε χρηματοπιστωτικό επίπεδο, κυρίως όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις ε, και τις αποζημιώσεις. Και αυτό είναι αδιαμπισβήτητα λάθος. Δεν μπορούμε μετά από κάποια χρόνια να επανέλθουμε στους πολίτες όταν ε, θα έχει προκύψει η επόμενη κρίση. Γιατί πολλοί έλεγαν ότι τέτοια γεγονότα ε, λαμβάνουν χώρα κάθε 100 χρόνια. Όχι όμως, τελικά ε, επαναλαμβάνονται κάθε 10 χρόνια. Έχουμε χάσει λοιπόν δυναμισμό, πρέπει να τον ανακτήσουμε. Και όλοι ε, εμείς που ε, συμμετέχουμε στη διαχείριση κρίσεων μετά τη Lehman Brothers δεν θα επανέλθουμε ποτέ σε αυτό που υπήρχε πριν από τη Lehman Brothers. Άρα δηλαδή πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε ε, θέματα που αφορούν ε, τους συστημικά τους θεσμούς, σε θέματα που αφορούν τα παράγωγα, σε μη συνεργάσιμες ε, δικαιοδοσίες και αυτό που έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία πρέπει να ασχοληθούμε με το σκιώδες ε, τραπεζικό σύστημα. Με κάποιους κατά προσέγγιση υπολογισμού της ΕΚΤΑ μιλάμε για το 35 μέχρι 40% του παγκόσμιου χρηματοψηφιακού συστήματος. Αυτό είναι το θέμα που χρήζει ρυθμίσεων. Αν θέλετε μπορώ ε, να αναφερθώ σε όλη την ατζέντα μεταρρυθμίσεων που είναι απαραίτητε να λάβουν χώρα στον χρηματοψηφιακό τομέα. Ε, μπορώ να σταματήσω εδώ, είμαι βεβαίω στη διάθεσή σα. Σίγουρα θα υπάρξουν και άλλε ερωτήσει. Μπορούμε να τη ρευνήσουμε περαιτέρω. σω να μην υπάρξει, να έχουμε χρόνο. Άλτε. Τώρα σωστή, σωστά βρήκα το όνομα. Τελικά το επόμενο μιλητή στον κατάλογο. Ε, Μια ερώτηση να κάνω για την επικοινωνία, λέει η κυρία Γκούλα, στα γερμανικά. Γι' αυτό ε, μιλήσατε ε, για κάτι ότι δεν έχει εναλλακτική λύση. Καταλαβαίνω τι λέτε. Δεν υπάρχουν τόσα όργανα παγκόσμια. Αλλά το 2010 αυτή η έκφραση είχε χαρακτηριστεί ως η δυσμενέστερη της χρονιάς ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση. Δεν μπορούμε να δίνουμε στους πολίτες ε, την αίσθηση ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος, γιατί δεν υπάρχει και χώρος για συζήτηση πλέον. Και ε, έχετε πει και στις ομιλίες σας ότι σας ενδιαφέρει πολύ η επικοινωνία με τους πολίτες και το πιστεύω. Αλλά όταν λέτε ότι χάσαμε την ευκαιρία κτλ. Είστε βέβαιος ότι η δημοκρατική νομιμότητα δεν χρειάζεται και λίγο χρόνο, δεν αξίζει και λίγο χρόνο. Γιατί δεν έχουμε προχώρησει τόσο πολύ. Επειδή πιστεύουν οι κυβερνήσεις ότι μπορούν να αποφασίζουν τα πάντα στο G20 ή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δηλαδή και μετά από μένα το χάος, δηλαδή. Ε, ε, μιλάω πάντα αγγλικά σε τέτοια φόρα, αλλά όταν κάποιος μιλάει τόσο θαυμάσια γερμανικά θα απαντήσω γερμανικά. Βεβαίως, ε, με συλλάβατε επ' αυτοφόρο, χρησιμοποιώ τη λέξη alternative loss, ότι δεν υπάρχει ανακτική λύση που στη Γερμανία όντως έτσι είχε χαρακτηριστεί το 2010. Δεν μιλώ για το περιεχόμενο των αποφάσεων, αλλά για την ύπαρξη του G20, που πραγματικά το θεωρώ εντάξει δεν είναι ιδεώδης κόσμος τον G20 αλλά καλύτερο δεν έχουμε και καλά θα κάναμε να ε, τον αξιοποιούμε όσες δυσκολίες και αν ε, συνεπάγεται αυτό. Είπατε κάτι σημαντικό για το χρόνο ότι οι αγορές ως ένα υποσύστημα έχουν άλλο χρόνο και άλλη λογική από την πολιτική ως υποσύνολο υποσύστημα και νομίζω ότι θα παραμείνει αυτό. Οι αγορές λειτουργούν σε κλάσματα του δευτερολέπτου πολλές φορές. Ενώ η ε, εργασία ε, για τη δημοκρατική νομιμοποίηση χρειάζεται χρόνο, για να το πω έτσι. Χρειάζεται συζήτηση και καταστάσεις που δεν ε, ανταποκρίνονται σε κάποιες θεωρίες από ορισμένα εγχειρίδια ε, για το απόλυτο της ε, αποτελεσματικότητας. Είμαστε πιο αργοί, αλλά πόσο πιο αργοί μπορούμε να είμαστε. Νομίζω σήμερα είμαστε υπερβολικά αργοί. Ε, δηλαδή αυτό που θα πρέπει να κάνουμε όχι να κοιτάμε στις οθόνες το Bloomberg και το Reuters πώς παίζουν οι διακοιμάνσεις με άγχος ε, το θέμα είναι να έχουμε ένα ε, στόχο προς τα που πηγαίνουμε και που θέλουμε να ε, στραφούμε. Και εδώ τίθεται ακριβώ το σωστό ερώτημα για τη δημοκρατική νομιμότητα. Μέχρι σήμερα, ειλικρινά, δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο δεν υπάρχει αντίστοιχη κοινοβουλευτική συνέλευση απέναντι στο G20. Θα μπορούσα, γιατί ε, την παραμονή συναντώνται 20 εργοδότες και 20 εργαζόμενοι ως συνδικάτα. Ε, τα 20 κοινοβούλια που είναι, δεν τα έχω δει ακόμα, δεν καταλαβαίνω γιατί. Λοιπόν, χρειάζεται υποστήριξη όντω για τα όσα πράττουμε, αλλά αυτό αφορά δύσκολα σημεία αναγκαστικά το ακούσαμε και το συζητήσαμε στην οικονομική διακυβέρνηση, θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Μετατοπίζεται η ευθύνη, εκχωρείται από τα εθνικά κοινοβούλια στο ευρωπαϊκό. Αυτό το θεωρώ λογικό βήμα, αλλά ορισμένοι δεν συμφωνούν πάρα πολύ. Είναι μια απαραίτητη συζήτηση που πρέπει οπωσδήποτε να γίνει και εσείς να την κάνετε βέβαια, δεν συμμετέχω σε αυτή. Εάν ε, όλα μπορούτε να τα κάνετε ε, στο Κοινοβούλιο ε, ή να ακολουθήσετε και το Συμβούλιο και να έχετε ένα είδος Κοινοβουλίου Ευρωζώνης. Αυτό είναι δικό σας θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Από τους συντηρητικούς, ο Ιβος Στρέζακ και πάλι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Άσμουσεν, έχω ερώτημα που βασίζεται σε ανοιχτές και αξιόπιστες πηγές Frankfurter Allgemeine Zeitung και Deutsche Presse. Και θέλω τα σχόλιά σας. Σχετικά με τη συνέντευξη του κυρίου Στόιμπλε για την Φραγκφούρτερ. Είπε λοιπόν ότι ε, Ίσως να χρειάζεται κούρεμα για τα ελληνικά ομόλογα. Μεγαλύτερο. Και η DPA ανέφερε ότι η γερμανική κυβέρνηση εξετάζει ένα σχέδιο που συνεπάγεται ένα κούρεμα 60% του ελληνικού χρέους. Σχόλιά σας σχετικά με αυτές τις ε, δύο σημαντικές πληροφορίες που σας παρουσίασα. Απάντηση. Είμαι πρόθυμος να σχολιάσω τις θέσεις του, της γερμανικής κυβερνήσεως. Αν τα πράγματα πάνε καλά δεν θα το κάνω αυτό στο μέλλον. Θα σχολιάσω τώρα. Στο μέλλον θα έχω διαφορετική τοποθέτηση όσον αφορά αυτό το θέμα. Εστε βέβαιος. Ο υπουργός μου είπε σε αυτή τη συνέντευξη ότι πρέπει να δούμε τι συμφωνήθηκε στις 21 Ιουλίου από του αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Ποιες λύσεις προτάθηκαν και να δούμε κατά πόσο οι προϋποθέσεις για τη συμφωνία που έλαβε χώρα εκεί εξακολουθούν να υπάρχουν. Αναφέρθηκε πιο συγκεκριμένα στην εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα για τα ελληνικά ομόλογα. Δεν αμφισβήτησε καθόλου την χρήση νέων μέσων για το EFSF. Αυτό χρειάζεται και χρειάζεται και γρήγορα. Βασιζόμαστε σε αυτά που συμβαίνουν στη Μάλτα και στη Σλοβακία σχετικά με το θέμα. Από εάν πρέπει τελικά να επιτευθεί ο φορολογικός στόχος, ο οικονομικός στόχος μάλλον, δηλαδή βιώσιμο χρέος για την Ελλάδα, αυτός είναι ο στόχος. Και πηγαίνουν προς τα πίσω. Η απώλεια του 21% που συμφωνήθηκε τον Ιούλιο ε, εξακολουθεί να ισχύει σαν στόχος. Αρκεί. Κύπας, περιμένουμε την ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους, της Τρόικα, που είναι κομμάτι της εκθέσεως συμμόρφωσης, να υποβάλει αυτά τα πορίσματα η Τρόικα και να δούμε που βρισκόμαστε και να συναγάγουμε τα αναγκαία συμπεράσματα. Πριν το κάνουμε αυτό, χρειάζονται συστήματα προστασίας, τύχη να ακολουθηθεί σωστή σειρά των κινήσεων χρειάζεται τάξη για τη χρηματοδοτική αγορά. Να αποφευθεί μια κάποια, κάποιο ε, γεγονός χρεοκοπίας ή κάτι συγκρίσιμο. Και είδα τις εκθέσεις του, που ακούστηκαν για κάποιο στοιχείο για κάποιο κούρεμα που χρειάζεται. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω ακόμα γιατί είναι στην Αθήνα ακόμα η Τρόικα. Αλλά δεν υπάρχει ακόμα αυτή η έκθεση βιωσιμότητας. Πρέπει να δούμε τι χρειάζεται να γίνει για να καταλήξουμε σε, βιολογι... σε βιώσιμη οικονομική κατάσταση μακροπρόθεσμα για την εν λόγω χώρα. Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω κανένα στοιχείο διότι δεν έχουμε μπροστά μας τα διάφορα μοντέλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τους πρασίνους, ο Σφέν. Αξιότιμα κυρία Άσμουσεν. Αναμφισβήτητα, εσείς είσαστε το πρόσωπο κλειδί της ε, χρηματοψηφιακής πολιτικής της Γερμανίας και ως πράσινος, ε, εγώ ε, πρέπει να σας πω ότι ξέρουμε ότι υπό τον κινθιανό flashback δουλέψατε ε, υπό τον ε, μεγάλο συνασπισμό, δουλέψατε ή σπουδάσατε στον κύριο Βάγγελ, στον κύριο Βέιμπα. Ε, έχετε λοιπόν ένα φάσμα γνώσεων και σπουδών και επιβιώσατε πολλών. Πριν από την κρίση είδαμε ένα ενδιαφέρον άρθρο για μεγαλύτερη απελευθέρωση της αγοράς χρεογράφων είδαμε ότι υπήρξε μια πρωτοβουλία που επιθυμεί να επιτύχει την απελευθέρωση της ε, ΙΚΑΜΠΕ, κάτι που απέτυχε και κατόπιν είδαμε ότι παίξατε και καθοριστικό ρόλο στην ε, κρίση τραπεζών, κάτι που κατά την άποψή μου στη Γερμανία δεν ε, συζητήθηκε διεξοδικά και απαρκώς. Εμείς έχουμε κάνει πολύ καλή εμπειρία με εσά, εμπειρία στην ομοθεσία, στα, στις τα κοινοβουλευτικά briefing ε, στην Ομοσπονδιακή Βουλή, στο Bundestag και πρέπει να πούμε ότι χαιρόμαστε που στο μέλλον ε, θα έχουμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, ε, έναν ρεαλιστή και όχι έναν δογματικό εμπειρογνώμονα. Θέλω λοιπόν να πω και να ρωτήσω το εξή. Ε, εφόσον πλέον δεν θα έχετε να δουλέψετε με διάφορου υπουργού, θα είσαστε σε έναν ανεξάρτητο θεσμό. Πώ θα συμπεριφερθείτε όταν η Τρόικα θα θελήσει να επιβάλλει όρους σε κράτη. Εμείς ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήταν ανέκαθεν εκείνος ο θεσμός που επιθυμούσε να επιβάλλονται σκληρά μέτρα και δεν λάμβανε παρκώς υπόψη του την κοινωνική διάσταση των προβλημάτων ούτε στην Ισπανία, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Ιρλανδία. Εσείς λοιπόν πώς θα προσπαθήσετε να ε, φέρετε και κάποια ισορροπία στα μέτρα που θα προτείνετε έτσι ώστε να μην αγνοηθεί πλήρως η κοινωνική διάσταση των προβλημάτων. Αξιότιμε κύριε Βουλευτά, Θα ήθελα και εγώ στο, να απαντήσω, να σχολιάσω το πρώτο σκέλος των παρατηρήσεών σας χωρίς ε, να αναφερθώ σε αυτό το άρθρο του 2006 ε, σχετικά με την τιτλοποίηση των χρεογράφων. Θα κάνω λοιπόν μία ανακεφαλαίωση. Και θα πω το εξή: Όλοι όσοι συμμετείχαν στη συζητήση τα τελευταία χρόνια για τη διαχείριση των κρίσεων, όλοι αναγκάστηκαν να νεοθεωρήσουν και να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Αυτό ισχύει και για μένα. Γιατί αυτή είναι μια χρηματοψητική κρίση που κανείς δεν την είχε προβλέψει ε, και γι' αυτό λοιπόν ε, αν κάποιος δεν αναθεωρεί την άποψή του σημαίνει ότι είναι ανεπίδεκτος μαθήσεως. Και εγώ δεν θέλω τουλάχιστον για τον εαυτό μου να ισχυριστώ ή να θεωρήσω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Η εμπειρία λοιπόν που συγκεντρώσαμε οδήγησε ε, στο ότι η τυφλή εμπιστοσύνη στην αγορά είναι, οδηγεί ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα όπως και ε, ο τυφλός δογματισμός. Εκείνο που χρειαζόμαστε είναι μια κοινωνία κρατών υπερεθνικούς θεσμούς έτσι ώστε να λαμβάνουν και κυρίως να εφαρμόζουν μέτρα. Το δεύτερο είναι σημαντικότερο. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Δεν νομίζω ότι ε, πρέπει να παρατηθούμε. Πράγματι, ε, χάσαμε κάτι από το δυναμισμό μας. Ε, αυτό το ρώτησε ο κύριος Μπούλμαν. Και δεν πρέπει να συμβεί το ίδιο, κυρίως στη Συμφωνία Βασιλεία 3. Νομίζω το χρωστάμε, το χρωστάμε να δείξουμε ότι βγάλαμε τα συμπεράσματά μας και μάθαμε. Όσον αφορά τώρα το συγκεκριμένο σας ερώτημα, δηλαδή στο μέλλον, πώς ακριβώς θα συμπεριφερθούμε. Εσείς ε, τάσεστε υπέρ του ρεαλιστή. Ξέρετε ότι στη Γερμανία ε, η λέξη ρεαλιστής ε, δεν είναι και τόσο ευπρόσδεκτη. Έβυχη μάλιστα, μάλλον έβυχη σε χρηματοπιστωτικό πλαίσιο όσον αφορά την αξία του χρήματος. Νομίζω όμως ότι και οι Γερμανοί πρέπει να μάθουν. Υπάρχουν άνθρωποι για τους οποίους τα επιτόκια είναι πάντα πολύ χαμηλά, άλλοι πάλι για τους οποίους τα επιτόκια είναι πάντα πολύ ψηλά. Λάθος και τα δύο. Πρέπει να δει κανείς ε, τα στοιχεία, τι συμβαίνει και από εκεί να εξάγει τα συμπεράσματά του. Η εμπειρική εργασία είναι πάντα το σημείο εκκίνησης για οποιοδήποτε θέση παίρνει κανείς με στόχο να επιτύχει τη σταθερότητα των τιμών. Όσον αφορά τώρα στη συγκεκριμένη θέση της ε, Τρόικα ή σε σχέση με την Τρόικα. Και εγώ πράγματι πιστεύω ότι στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται να είναι κανείς σκληρός. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η σκληρότητα ισούται με την ε, κοινωνική ψυχρότητα, γιατί σε τελική ανάλυση τίποτα δεν είναι πιο αντικοινωνικό από το να μην υπάρχει ένας εφαρμόσιμος ή εκτελεστέος προϋπολογισμός. Τίποτα δεν είναι πιο αντικοινωνικό από τον υψηλό πληθωρισμό. Νομίζω γνωρίζετε όλοι σας ε, το ε, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει και αυτό εξάγει τα συμπεράσματά του από την Ασία και νομίζω κατόπιν τούτου ε, αυτό ε, θα το βοηθήσει να αντιμετωπίσει καλύτερα την κατάσταση στην Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία. Ε, θα ήθελα να πω ότι πέντε λεπτά κανονικά θα έπρεπε να ισχύει η ερωταπάντηση. Μέχρι τώρα το έχουμε ξεπεράσει. Πάω στους πράσινους. Ε, θα έχουμε τέσσερα λεπτά για την ερώτηση, στη, στην ΚΟΕ με συγχωρείτε, στην ΚΟΕ, στην αριστερά. Ε, θα πρέπει να έχουμε τέσσερα λεπτά, αλλιώς ε, αργότερα θα αναγκαστούμε να περιορίσουμε τον χρόνο. Ο Γιούργεν έχει το λόγο. Εκτός μικροφώνου ο Γιούργεν, δυστυχώς. Στο μικρόφωνο παρακαλώ. Ευχαριστώ. Τώρα ακούγεται. Κύριε Άσμουσεν, όπω πολύ καλά γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόσφατα ενέκρινε το πακέτο για την οικονομική διακυβέρνηση. Και αυτό ε, στο πλαίσιο τη επιτήρηση των δημοσιονομικών εκτροχιασμών έχουμε πλεονάσματα στι εξαγωγέ. Αυτό ισχύει για τη Γερμανία εδώ και χρόνια και αυτό είναι προβληματικό. Οικονομολόγοι όπω ο Χάνε Φλάσπεκ ε, θεωρούν ότι αυτό είναι και ένα από τα βασικά αίτια που προκάλεσε την κρίση. Βέβαια η γερμανική κυβέρνηση τάσεται κατά αυτής της μονόπλευρης ε, θεώρησης των πραγμάτων και προσπαθεί να αγνοήσει και να παραγωνίσει αυτό το στοιχείο των εμπορικών πλεονασμάτων. Ερωτώ λοιπόν εσάς, εσείς ε, αυτά που συζητήσαμε εδώ στην Επιτροπή μας και στο Κοινοβούλιο τα συμμερίζεστε και κατά την άποψή σας οι μεγάλες ε, οικονομίες της Ευρωζώνης που έχουν μεγάλα εμπορικά ελλείμματα πώς πρέπει να συμβάλλουν για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι ανισορροπίες. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Και η δεύτερη μου ερώτηση είναι η Σε διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συσσωρεύονται αντιδράσεις ε, κυρίω των νέων που πλήττονται από τα μέτρα λιτότητας. Εμένα με ενδιαφέρει ποια είναι η δική σα απόφαση και τι ρόλο θα παίξουν αυτέ οι διαμαρτυρίες στι πολιτικέ αποφάσει που θα κληθείτε να λάβετε. Απάντηση. Ε, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος όπως μου επισημάντηκε. Πράγματι, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό μακροοικονομικές ανισορροπίες στο τέλος να λαμβάνονται υπόψη σε αυτή τη διαδικασία επιτήρησης. Γιατί αυτό πράγματι μέχρι τώρα ήταν μία μαύρη κοιλίδα στο σύμφωνο σταθερότητας ε, και το γεγονός ότι προέκυψαν ανισορροπίες ε, αυτό ε, οδήγησε στην κρίση που μαστίζει ορισμένα Στο πλαίσιο της διαδικασίας λοιπόν επιτήρησης, ανισορροπίες ε, που εκφράζονται είτε με δημοσιονομικά ελλείμματα είτε με εμπορικά πλεονάσματα, όλα αυτά θα παρακολουθούνται, αλλά πράγματι εδώ έχουμε μια ασύμετρη στάση και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε βάρος κυρίως σε τομείς που παρουσιάζουν ελλείμματα, κυρίως σε θέματα ανταγωνιστικότητας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι και τα κράτη δεν πρέπει να κάνουν τίποτα. Όχι. Ε, τα κράτη πρέπει να στηρίξουν την εσωτερική τους ζήτηση να εφαρμόσουν ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Εγώ προσπάθησα να σα δώσω τι απαντήσει μου γραπτά. Δηλαδή μιλάω για την αγορά παροχή υπηρεσιών, για την παιδεία, για την έρευνα και την ανάπτυξη, ε, την αγορά εργασία ε, και γραπτά καθιστώ με απόλυτη σαφήνεια πώς εγώ ορίζω την αγορά ή την εργασία Επίσης εσείς ρωτήσατε ή τοποθετηθήκατε στις διαμαρτυρίες, στους αγανακτισμένους όπως λέμε, σε ορισμένα κράτη-μέλη ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης κυρίως. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι ένα καμπανάκι, θα το χαρακτήριζα. Καμπανάκι για όλους εκείνους που ασχολούνται με την πολιτική. 45% είναι η ανεργία των νέων στην Ισπανία. Και αν το λίγα εκεί, βλέποντας μάλλον κανείς ε, τις εικόνες, τηλεόραση, είναι νέοι σαν και εμένα. Είναι λοιπόν ένα καμπανάκι που σωστά ηχεί κατόπιν τούτου το θέμα εκπαιδευτικά συστήματα είναι καθοριστική σημασία. Η πρόσβαση στην εκπαίδευση είναι πολύ σημαντικό. Εμένα η μητέρα μου ήταν δασκάλα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό όλοι να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην παιδεία, ξεκινώντα από τον υπηαγωγείο, να έχουν όλοι πρόσβαση σε όλε τι ε, κλίμακε τη παιδείας και μέσω ε, κρατικών ενισχύσεων. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα από το Λαϊκό Κόμμα, ο Βερναλάγκεν. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Άσμουσεν. Ε, ε, για το βιογραφικό σας, εγώ δεν αμφισβητώ τίποτα. Ε, δεν χρειαζόμαστε τέτοια κηρύγματα τύπου Γκίγκολτ. Ξέρουμε ότι είστε ειδικό η ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής ε, Τράπεζας αφισβητήθηκε ακριβώς επειδή εξαγόρασε ε, τα κρατικά ομόλογα. Θέλω την άποψή σας γι' αυτό. Στη συνέχεια για το FSF μας είπατε ότι χρειάζονται νέα μέσα και εργαλεία. Ο κύριος ε, Τρισέ απέριψε τις άδειες των τραπεζών και την επανακεφαλαιοποίηση. Αυτό πώς θα γίνει τότε και η στόχη της ΕΚΤ τρίτο σήμερα επικεντρώνεται στη σταθερότητα των τιμών και προσεχώς και στη σταθερότητα των χρηματαγορών. Και τι λέτε για αυτά που προτείνει η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, αναζωογόνηση της οικονομικής δραστηριότητας. Και να πω κάτι σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Μπούλμαν, για το σύμφωνο σταθερότητα, συχνά τα κράτη-μέλη μπλόκαραν την νομοθεσία. Τώρα το σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη ε, είτε πρόκειται για το 2003 που ήσασταν εσεί στο Υπουργείο Οικονομικών ήδη, είτε πρόκειται για την κοινωνική μέθοδο που σήμερα έχει πέσει σε λύθη ή ε, συγκεκριμένοι στόχοι των κρατών μελών τα οποία μπλοκάρονται εκεί στο ΕΜΙΑ που αναφέρετε κι εσείς. Τι γίνεται λοιπόν ε, με τη ρύθμιση των χρηματαγορών και ε, πού θα είχατε δεχομένως προτάσεις να κάνετε. Μας συστήσατε να δημιουργήσουμε ένα κοινοβούλιο των G20, θαυμάσια ιδέα. Αλλά μήπως αρκεί ε, η κοινοτική μέθοδος να λάβει απλούστατα πιο σοβαρά υπόψη της το υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οχτώ ερωτήσεις κάνατε κύριε Λάγκεν μου. Θα προσπαθήσω ε, γρήγορα να απαντήσω. Ε, ρωτήσατε για την ανεξαρτησία της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε σχέση με το συγκεκριμένο πρόγραμμα που ακολουθήσαμε τελευταία. η ανεξαρτησία μιας κεντρικής τράπεζας είναι υποχρεωτική και αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς πλέον σε ένα σύγχρονο οικονομικό παγκόσμιο σύστημα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η ανεξαρτησία και η λογοδοσία δεν είναι διόψεις του ίδιου νομίσματος. Είναι αλληλένδετα. Οι αποφάσεις για ε, το τελευταίο σύστημα ε, για την εξαγορά των ομολόγων ε, δεν διακυβεύουν την αξιοπιστία και την ανεξαρτησία της τράπεζας. Ο νομισματικός μηχανισμός ε, διακίνησης ε, είχε διακυβευτεί, είχε διαταραχθεί, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα κρατικά ομόλογα, που παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο για άλλα τμήματα της εθνικής οικονομίας. Γι' αυτό το έκανε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στα πλαίσια της εντολής της. Για μένα όμως είναι σημαντικό να είναι περιορισμένο χρονικά αυτό, και σε όγκο και να είναι τέλεια η αποστήρωση αυτών των ε, δράσεων για να μην ε, υπάρχει πίεση στην ε, σταθερότητα των τιμών. Για το EFSF νομίζω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να έρθουν και γρήγορα τα τέσσερα νέα μέσα αγορές. στην πρωτογενή αγορά, στη δευτερογενή αγορά έχει πολύ σημαντικό ρόλο αυτό για να μπορεί ο FSF να δραστηριοποιείται στη δευτερογενή αγορά. Τρίτον, επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών μέσω τη κεντρική κυβέρνηση, εκάστοτε. Και το τέταρτο, ένα λεγόμενο ε, ε, προφυλακτικό μέσο, precautionary instrument, για να μην έχουμε ε, κίνδυνο διασποράς του φαινομένου. Θα πρέπει να είναι συγκεκριμένος και ο όγκος του ΕΦΣΕΦ χωρίς πρόσβαση όμως ε, στη ρευστότητα της Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Γιατί αυτό αντιτίθεται και στο πνεύμα και ε, στο γράμμα της συνθήκης και συγκεκριμένα στο άρθρο 123. Ε, με ρωτάτε αν θα είχε νόημα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να καταρτήσει ένα κατάλογο στόχων όπως έχει η ομόλογη τράπεζα στις Ηνωμένε Πολιτείες με ισότιμους στόχους και πολλαπλούς έχει η ΦΕΤ. Αυτό το ερώτημα δεν τίθεται για μένα. Η συνθήκη ορίζει ε, την εντολή της τράπεζας. Είναι σωστό αυτό, βασίζεται στις ε, παραδόσεις ολόκληρης της Ευρώπης και αυτό τώρα θα πρέπει να εφαρμόσουμε λογικά στην πράξη. Άλλη ερώτηση. Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και το άλλο οι χρηματαγορές και η ρύθμισή τους. Είναι επίσης εκ των όνου κάνευ. Είτε πρόκειται τώρα για το δημοσιονομικό συντονισμό ή τη ρύθμιση των χρηματαγορών, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει αυτό που ονομάζουν στα αγγλικά ownership. Θα πρέπει να κάνουν κτήμα τους ε, ε, αυτό το εγχείρημα. Πιο στενή δηλαδή ε, δημοσιονομική συνεννόηση ε, αλλά αυτό αφορά και τη ρύθμιση των χρηματαγορών. Υπάρχει μια διαφορά εκεί στις χρηματαγορές. Αυτό είναι θέμα της εσωτερικής αγοράς, δηλαδή και των 27 κρατών. Αλλά το δημοσιονομικό υπάρχουν ε, εύλογοι ε, λόγοι να συνεργαστούν περισσότερο οι χώρες της Νομισματικής Ένωσης για να γίνει πιο δυνατή, πιο ισχυρή. Για μένα έχει μεγάλη σημασία αυτό. Όσα μπορούμε να τα υλοποιούμε σε επίπεδο 27, αλλά τα θέματα που έχουν να κάνουν με το κοινό νόμισμα μπορούν να γίνουν και σε επίπεδο 17. Η 17 είναι μια κλειστή λέσχη. Το έδειξε αυτό και η ένταξη της Εσθονίας σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Τα κριτήρια σύγκλησης είναι ένα θέμα και όταν κάποιοι τα πληρούν ε, ε, πάγια και σωστά και σταθερά ε, μπορούν να ενταχθούν στην νομισματική ένωση. Αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν και στην κοινοτική μέθοδο είναι οι κυβερνήσεις να εστερνίζονται αυτή την προσπάθεια και όχι μόνο οι κυβερνήσεις αλλά και τα κοινοβούλια των μεμονωμένων κρατών μελών. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα ο Ντολίν Σάντσες Πρεσέδο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Άσμουσεν, Εκτιμώ πάρα πολύ την εμπειρία σας και τη σαφήνεια των απαντήσεών σας. Ιδιαίτερα τη θέση σας υπέρ του φόρου χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Είναι ένα θέμα ε, που ε, ε, αφορά και την Κεντρική Τράπεζα. Το θέμα της σταθερότητας των τιμών και των δύστιχου στόχου. Θεωρείτε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν κίνδυνοι πληθωρισμού πήγε αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας στις ΗΠΑ και εκεί θεωρούν ότι ο κίνδυνος είναι ο απόπληθωρισμός και τα χαμηλά επιτόκια θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε λύση των προβλημάτων του χρέους και σε τόνωση της ανάπτυξης. Θα μπορούσε να υπάρξει ένα σενάριο με χαμηλά επιτόκια όπως είναι οι Ηνωμένε και άλλες πολιτικές, κοινωνικός διάλογος, άλλες δημοσιονομικές πολιτικές εκτός από τη νομισματική με ένα οικονομικό, ε, δημοσιονομικό και νομισματικό ε, μείγμα. Και η Κεντρική Τράπεζα και το EFSF ε, ή ο μελλοντικός μηχανισμός ESM θεωρείται ότι δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν με άμεσο τρόπο. Και πώς θα βρεθούν οι απαρκείς και απαραίτητοι πόροι από άλλες πηγές. Ελπίζω ότι ερμηνεύω σωστά το ερώτημά σας. Ε, αν ακολουθήσω λάθος κατεύθυνση μπορείτε να διαμαρτυρηθείτε αν δεν σας δώσω σωστέ απαντήσει. Το ερώτημά σας λοιπόν είναι ποια είναι η προοπτική όσον αφορά τον πληθωρισμό. Από εκεί ξεκινήσατε. Εγώ θα έλεγα ότι τα στοιχεία του πληθωρισμού που ήταν περίπου 3% στα στοιχεία που εκδόθηκαν για την Ευρωζώνη. Είναι σαφώ πάνω από το στόχο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δηλαδή ότι ένα επίπεδο πληθωρισμού που οδηγεί στη σταθερότητα τιμών. Πιθανότατα θα παραμείνει πάνω από το 2% για κάποιους μήνες, αλλά ίσως τελικά επιστρέψουμε στο πεδίο του 2%. Κάτι που θα ευθυγραμμίζεται με σταθερότητα των τιμών μεσοπρόθεσμα μπορούμε να πούμε ότι οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό, από τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη είναι ισορροπημένοι. Βλέποντας πού βρισκόμαστε τώρα. Ρωτήσατε μετά το πολιτικό μείγμα στην Ευρωζώνη ή στις ΗΠΑ. Λαμβάνοντας υπόψη την ότι η ΕΚΤ και η ΦΕΔ έχουν διαφορετική εντολή, εντελώς διαφορετική. Αυτό το ανέφερα. 100% έχετε δίκιο. Σημαντικό είναι το πολιτικό κράμα, ε, το κράμα των πολιτικών που εφαρμόζεται σε μακροοικονομικό επίπεδο και μικροοικονομικό. Εδώ η ΕΚΤ έχει περιορισμένη αλλά σημαντική εντολή ταυτόχρονα. Πρωταρχικά να πετύχει σταθερότητα τιμών. Α, εκεί μπορεί να συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι κυβερνήσεις μετά, κυρίως σε επίπεδο κρατών μελών, μέσω εργαλείων όπως η φορολογική πολιτική ή διαθωτικές πολιτικές στην ευρύτερη με την ευρύτερη έννοια του όρου συμβάλλουν στο δυναμικό ανάπτυξης της οικονομίας, στον καθορισμό των αμοιβών, κάτι που διοργανώνεται μέσω συμφωνιών μεταξύ εργοδοτών και συνδικάτων σε περισσότερες, περισσότερες χώρες, σύμφωνα με κανόνες μισθοδοσίας και αμοιβών στην Ευρώπη, Όλοι πρέπει να συμβάλλουν, ο καθένας στα πλαίσια ευθυνών του. Δεν θα πρέπει να ανακατευθούν αυτές οι αρμοδιότητες. Γι' αυτό σημαίνω ότι το άρθρο 123 της συνθήκης είναι πολύ κρίσιμο. Άρθρο που απαγορεύει την νομισματική χρηματοδότηση της φορολογίας. Είναι το πνεύμα που πρέπει να ακολουθήσουμε του κειμένου. Χρειαζόμαστε διαχωρισμό. Τι κάνει η νομισματική πολιτική, ποια είναι η εντολή που έχει δοθεί και η οικονομική, η φορολογική. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Το άρθρο αυτό είναι από τους βασικούς πυλώνες του, του πλαισίου για τη νομισματική πολιτική στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλοι Σμιτ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Άσμουσεν, ήσασταν στο επίκεντρο κάθε καταιγίδα ε, τελευταία χρόνια και από τους βασικούς ε, πρωταγωνιστές στη Γερμανία. Και η Γερμανία φέρει και ιδιαίτερη ευθύνη και υποχρέωση στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στην Ευρωζώνη θα λέγατε ότι η γερμανική ηγεσία ανέλαβε τις ευθύνες της κατά τη διάρκεια των ετών αυτών. Και δεύτερη ερώτηση αφορά το εξή. Εγώ είμαι Σουηδός, εκτός Ευρωζώνης δηλαδή η χώρα μου. Θα είχε νόημα, θα συμβουλεύατε τώρα να μπουν στο ευρώ με την κατάσταση που ισχύει αυτό τον καιρό και νέες χώρες. Θα ήσασταν υπέρ για τη χώρα όμω που αν μπορώ να σας ρωτήσω, είστε υπέρ της ένταξη τη Σουηδίας αυτή τη στιγμή στην Ευρωζώνη. On your first... Στην πρώτη σας ερώτηση, κατά πόσο η γερμανική ηγεσία έπραξε τα δέοντα κατά τη διάρκεια της κρίσης, η απάντηση είναι καταφατική. Να σας πω ποιο θα μπορούσε να ε, είναι το κριτήριο που θα με καθοδηγεί ε, στο μέλλον, αν με ορίσετε. Δεν πρόκειται ποτέ να επικρίνω καμία κυβέρνηση, ούτε το γερμανική ούτε καμία άλλη, για αποφάσεις που έλαβαν στο παρελθόν όσο ήμουν εγώ δημόσιος υπάλληλο κρατικός λειτουργός για τη γερμανική κυβέρνηση. Στο μέλλον μπορεί να αλλάξει ε, πολύ διαφορετικά να είναι η θεώρηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι πιστό στο σημερινό μου εργοδότη να κοιτάξω το παρελθόν και να πω ότι αυτά που κάνατε στο παρελθόν ήταν λάθο. Θα κάνω μια σαφή διάκριση. Ο γέγονε γέγονε και από εδώ και πέρα είναι διαφορετικός ο ρόλος μου σε περίπτωση που θα αναλάβω. για την νομισματική ένωση. Ε, συναισθηματικά θα μπορούσα να πω εγώ να μπω τον πειρασμό ότι μια χώρα με τέτοια παράδοση και πολιτιστική και δημοσιονομική, αν θέλετε να μπείτε στην Ευρωζώνη, καλώς να ορίσετε. Αλλά αυτή δεν είναι η απόφαση. Η, η Νομισματική Ένωση δεν είναι κλειστή λέσχη. Υπάρχουν κριτήρια, τέσσερα, θα πρέπει βιώσιμα και αηφόρα κάποιος να τα πλήρει, όχι για ένα-δύο χρόνια και τελείωσε. Όχι, θα πρέπει να είναι ε, τα στοιχεία σωστά και να ελέγχονται. Αυτό είναι ένα δίδαγμα του παρελθόντος. Και υπάρχουν και άλλες ευθύνες που ορίζει η συνθήκη ε, για το pre-in. Ε, μελλοντικές χώρες που ενδεχομένω να ενταχθούν θα πρέπει να περάσουν κάποια στάδια, είναι γνωστή η διαδικασία και καλώς έχει, αλλά ε, αυτή είναι η επίσημη απάντησή μου. Συναισθηματικά θα έτεινα να απαντήσω ότι η Σουηδία βεβαίω, εφόσον πληρεί τα κλειδίρια, θα είναι μια καλή χώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ευπρόσδεκτη. Αυτό δεν το λέω 100% επίσημα, αλλά το λέω με την καρδιά μου. Ναι, εγώ πιστεύω στο μέλλον τη Ευρωζώνης βεβαίω, Δεν τίθεται καν ε, θέμα σήμερα. Πριν από λίγου μήνε εντάχθηκε η Εστονία και έχω την αίσθηση ότι είναι ε, γενικά ικανοποιημένοι που συμμετέχουν στη Λέσχη, βεβαίω. Και η υποστήριξη για την Ευρώπη στην Εστονία στις δημοσκοπήσεις είναι πολύ ψηλότερη από ό,τι στη Γερμανία. Και όπως σας είπα στο παρελθόν υπάρχουν κριτήρια οικονομικά και νομισματικά που πρέπει κανείς να πληρεί. Αλλά αυτή τη στιγμή μπει κανείς στη λέσχη αυτή, ε, λαμβάνει μέρος της αποφάσης. Αυτό δεν θα πρέπει να το λησμονούμε ποτέ. Ευχαριστώ πολύ. Το ECR είπε ότι τελείωσε με τις ερωτήσεις που είχε να υποβάλει, οπότε επανερχόμαστε στους πράσινους. Βεν, αν έχεις κάτι άλλο να ρωτήσεις, αν θες. Ε. Θα ήθελα να αφήσω τους συναδέλφους να πάρουν το λόγο, αν είναι άλλοι που θέλουν να ρωτήσουν. Πρόεδρος, το ΕΛΚ νομίζω είπε ότι τελείωσαν τις ερωτήσεις του. Ναι. Οπότε έχουμε χρόνο αν θέλετε. Καλώς. Έχω άλλη μια ερώτηση. Έχω μπερδευτεί κάπως. Όσον αφορά τις απόψεις για την νομισματική πολιτική. Θα μπορούσατε να μας διαφωτίσετε. Κυρίως όσον αφορά ένα συγκεκριμένο θέμα που με έχει εκπλήξει από την κρίση. Ο ορισμός του πληθωρισμού βασίζεται κατά πολύ στον πληθωρισμό τιμών καταναλωτών. Αλλά είδαμε σημαντικά προβλήματα και στις ε, αγορές ε, στοιχείων ενεργητικού. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να αναπτύξει περισσότερο τον ορισμό της αθερότητας τιμών βλέποντας τη διακύμανση των ε, στοιχείων ενεργητικού, των τιμών των στοιχείων ενεργητικού, για να το πω έτσι γενικά. Όταν σας μπέρδευσα, σημαίνει ότι δεν έκανα ε, καλή δουλειά. Προσπάθησα να το πω στην εισαγωγική μου ομιλία είπα ότι οι φυσαλίδες στις χρηματιστικές αγορές ε, και στην αγορά κινήτων που τροφοδοτήθηκαν από, από τροφοδοσία σε χρήμα κλπ. δεν είχαν θεωρηθεί σαν τμήμα της νομισματικής πολιτικής. Είχα, στην αρχή προσπάθησα να πω τι έπρεπε να γίνει. Προσπάθησα να ξεκαθαρίσω περαιτέρω το όλο θέμα. Νομίζω ότι θα τηρούσα τον ορισμό της σταθερότητας των τιμών χρησιμοποιώντας τους εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτού. Είναι κάτι διαφανές, συγκρίσιμο, όχι μόνο στην Ένωση αλλά σε όλο τον κόσμο. Εάν χάσουμε αυτόν τον ορισμό, ίσως χάσουμε κάποια διαφάνεια που έχουμε πετύχει. Όμως, νομίζω, όπως είπα, ότι η πολιτική της αναμονής όσον αφορά το πληθωρισμό των τιμών προσαρμόστηκε, άλλαξε από το 2007-2008 όσον αφορά την νομισματική πολιτική και τις συζητήσεις που γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο και σωστά. Τώρα υποστηρίζουμε την προσέγγιση που πάει κόντρα στον άνεμο, αν θέλετε, όσον αφορά αυτό το θέμα, κόντρα στο ρεύμα. Το ερώτημα, το θέμα είναι ποια μέσα έχουμε στη διάθεσή μας. Γίνεται πολλή έρευνα. Πρέπει να γίνει έρευνα στον τομέα αυτό. Διότι όταν κολλούμε στις παλιές αρχές ότι όταν έχεις πάνω από ένα στόχο χρειάζεται θεωρητικά πάνω από ένα μέσο, αν έχεις ένα βασικό μέσο επιτόκια σαν κεντρική τράπεζα, έχεις στόχο τη σταθερότητα τιμών. Αν το κάνεις αυτό, ίσως να αντιμετωπίσεις δυσκολίες. Έχω περιορισμένες γνώσεις εδώ. Έχουμε περιορισμένες γνώσεις. Χρειάζεται έρευνα. Για κάποια εργαλεία για μακροοικονομική συνετή διαχείριση που ίσως θα μπορούσαν να αναπτυχθούν. Χρειάζεται, χρειάζεται στα, περιγράφεται στα κίνητα, χρειάζεται. Ε, αλλά για συγκεκριμένες λύσεις χρειάζεται πολλής δρόμος. Πρέπει να δούμε τον πληθωρισμό των στοιχείων ενεργητικού και ότι αυτός ο πληθωρισμός οδηγεί σε κινδύνους για σταθερότητα των τιμών. Αυτή η προσέγγιση είναι σωστή και κατά κάποιο τρόπο Πώ να το πω, δεν είναι αστείο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει δύο πυλώνε όσον αφορά το πλαίσιο που ακολουθεί για την νομισματική πολιτική. Αυτή η στατική των δύο πυλώνων εστιάζεται σε οικονομικέ πτυχέ και σε νομισματικέ πτυχέ. Και θεωρήθηκε προ κάποιων ετών ότι υπήρχε δίδεται μεγαλύτερη σημασία στον οικονομικό πυλώνα της νομισματικής στρατηγικής. Και τώρα Κινούμεθα περισσότερο προς την νομισματική πολιτική και τις σχετικές πτυχές που δεν υπάρχει ισορροπία πια στη στρατηγική των δύο πυλώνων. Ανάπτυξη και σώρευση χρημάτων και όγκοι πιστώσεων πρέπει να εξετάζονται όταν έχεις αυτού του είδους τον πληθωρισμό δηλαδή των διαφόρων στοιχείων του ενεργητικού στην τιμή των χρεογράφων. Ευχαριστώ πολύ. Η Ελίσσα. Θα μιλήσω πορτογαλικά αν δεν σας πειράζει. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας ε, σήμερα εδώ. Θα ήθελα λοιπόν να επανέλθω στην ε, απάντηση που δώσατε στο συνάδελφο κύριο Γκοζέ. Δηλαδή, στο ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα πακέτο παρεμβάσεων, κυρίως ε, έχω την εντύπωση ότι ζούμε σε μία περίοδο φαύλων κύκλων και θα εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ. Ε, θα θυμάστε ότι ήταν απαραίτητο και είναι απαραίτητο ε, να υπάρξει επανακεφαλοποίηση τραπεζών. Αυτή λοιπόν η επανακεφαλοποίηση ε, θα πρέπει να γίνει από πλευρά κρατών, όμως αυτή τη στιγμή πολλά κράτη αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν γιατί έχουν υπερβολικό έλλειμμα. Οι τράπεζες όμως εξακολουθούν να είναι οι μεσάζοντες χρηματοδότησης του δημόσιου χρέους. Άρα δηλαδή μιλάμε για ένα αρνητικό σπιράλ το οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή να πάυσει να υπάρχει. Αυτή τη στιγμή έχουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην οποία υπάρχει κάποιο, κάποια διαίρεση, διχασμός. Από τη μια ε, λένε ότι είναι, υπάρχουν τράπεζες που είναι υπερβολικά μεγάλες ε, για να ε, σωθούν και πολλά κράτη που είναι πολλά μεγάλα για να μη σωθούν. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Κατά τη δική μου άποψη οφείλουμε αφενός να ε, προχωρήσουμε με την ε, αντιμετώπιση των τραπεζικών κρίσεων. Η Κομισιόν πρότεινε νομοθετικό σχέδιο μέσα στο Νοέμβρη, αλλά κατά την άποψή μου ε, θα πρέπει να γίνει πιο γρήγορα. επίγει το θέμα. Κυρίως θα πρέπει να συμφωνήσουμε στο ότι οι τράπεζες οφείλουν να αυτοχρηματοδοτηθούν μόνες τους να σωθούν αντί να το παραπέμπουν κάπου αλλού. Κατά τα άλλα πρέπει να βρούμε τρόπους διαχείρισης δημοσίων χρεών για να αποφύγουμε επιμόλυνση που κατά την άποψή μου δεν θα προσφέρει τίποτα. Ε, οι τράπεζες ε, δεν μπορούμε να λέμε ε, χρηματοδοτήστε την ε, Ελλάδα και από την άλλη αυτά που δίνεται θα υποστούν κούρεμα της τάξης του 30% του 40%. Προφανώς εδώ κάτι δεν πάει καλά και αυτό πρέπει να διορθωθεί. Η κατάσταση σαφώς και είναι περίπλοκη. Θα ήθελα όμως να γνωρίζω από εσάς να μας πείτε ποια είναι ε, τα στοιχεία του πακέτου που οραματίζεστε. Ε, Μα είπατε κάποιε γενικέ αρχέ, αλλά ίσω μπορείτε να μπείτε σε περισσότερε λεπτομέρειε κυρίω να μα διευκρινίσετε ποιο ακριβώ θα είναι ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε όλο αυτό το πλαίσιο. No, Σας ευχαριστώ πολύ ε, για αυτή την ε, ερώτησή σας και συμφωνώ απόλυτα ότι μετά από 1,5 χρόνο όπου μένεται η κρίση στην Ευρωζώνη, κάτι πρέπει να αλλάξει, γιατί αλλιώς θα χάσουμε όλη την αξιοπιστία μας. Και έχετε απόλυτα δίκιο. Πρέπει να τερματίσουμε, να διακόψουμε αυτόν τον φαυλοκύκλο που προέρχεται από τη δημοσιονομική κατάσταση των κρατών, πάει στις τράπεζες, από τις τράπεζες περνάει στην πραγματική οικονομία ε, και μετά μέσα από ε, το φορολογικό σύστημα περνάει στα κράτη. Αυτός ο φαύλος κύκλος πρέπει να σπάσει. Η κατάσταση λοιπόν είναι η εξής. Κατά κάποιον τρόπο μοιάζει ε, στο 2008, από την άλλη όμως παράλληλα διαφέρει και πάρα πολύ από το 2008. Αυτό που είναι τελείως διαφορετικό είναι ότι το 2008 το πρόβλημα ξεκίνησε με την ποιότητα δραστηριοτήτων ορισμένων τραπεζών εκτός ισολογισμών και μετά οι ενέργειες αυτές πέρασαν στα ισοζύγια, στους ισολογισμούς με συγχωρείτε, των κρατών. Τα περίφημα ε, τοξικά προϊόντα. Τώρα όμως το πρόβλημα ξεκίνησε από τη δημοσιονομική κατάσταση ορισμένων κρατών. Δεν είναι πλέον δεδομένη η βιωσιμότητα δημόσιου χρέους. Πρέπει κανείς να την κερδίσει. Και αυτό σίγουρα έχει επιπτώσει στους ισολογισμούς των τραπεζών. Τώρα λοιπόν πρέπει η αντίδραση να ξεκινήσει από το κράτος και να περάσει στις τράπεζες. Και αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Προφανώς εκείνο που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να ισχυριζόμαστε ότι τα κρατικά χρόγραφα είναι τοξικά και ότι ε, πρέπει οι ε, ισολογισμοί των ε, κρατών να απελευθερωθούν από αυτά τα τοξικά προϊόντα. Δεν γίνεται αυτό. Ε, αυτό αποκλείεται. Πρέπει λοιπόν να βρούμε μια άλλη λύση σε σχέση με το 2008. Και για να είμαι σαφής, εγώ δεν θέλω να πω τίποτα για ποσοστά ή ενδεχόμενο ύψος ε, κουρέματο. Ε, δεν θέλω να αναφερθώ σε οτιδήποτε έχει σχέση με τη λύση του προβλήματος της Ελλάδας. Τώρα, όσον αφορά το πακέτο και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είπα ότι πρέπει να έχουμε ένα περιεκτικό πακέτο σύντομα, όσο πιο σύντομα γίνεται, διότι διαδίδεται η επιμόλυνση και αυτό το περιεκτικό πακέτο πρέπει να περιλαμβάνει πρώτον μια αξιόπιστη λύση για την Ελλάδα στο δημοσιονομικό επίπεδο, αλλά ακόμα περισσότερο στο θέμα της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Πρέπει να δούμε πώς μπορεί να σημειώσει ανάπτυξη η Ελλάδα. Η Ελλάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ο ανατολικότερος εταίρος της δύση. Ήταν η ανατολική κοινή πλευρά που μπορούσαν να γίνουν δουλειές, business, υπό την αιγύρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν γίνεται. Πρέπει να βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος. Δεύτερον, χρειαζόμαστε στεγανά στο πλαίσιο ενός διευρυμένου ε, μηχανισμού στήριξης, η FSF. Τρίτον, χρειαζόμαστε έναν τρόπο ε, που δεν θα προκαλεί στιγματισμό. Η ανακεφαλοποίηση των ευρωπαϊκών τραπεζών και παράλληλα η διασφάλιση των βραχυπρόθεσμων αναγκών τους χρηματοδότησης. Χρειαζόμαστε εξάλλου ε, αξιόπιστες ε, οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές, όχι μόνο σε ευρωπληματικές χώρες, αλλά και σε χώρες που ενδεχομένως να έχουν μολυνθεί ή να μολυνθούν από άλλες, ακόμα και μεγάλες χώρες προφανώς. Και πρέπει τέλος να ξεκαθαρίσουμε πού ακριβώς βαδίζουμε, πού βαδίζει η Ευρώπη. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια δομή διακυβέρνησης η οποία θα εστιάζεται ξεκάθαρα στην Ευρωζώνη. Και εάν όλα αυτά τα συνδυάσουμε μπορούμε τελικά να καταλήξουμε ε, σε γενικές κουβέντες, περισσότερη ενσωμάτωση, οικονομική διακυβέρνηση. Μα τι σημαίνουν ακριβώς όλα αυτά. Σημαίνουν ότι οι φτωχότερες χώρες θα πρέπει να πλέον περισσότερο και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τις ε, λιγότερο ε, από τις φτωχότερες, στις χώρες. Δεν μιλάμε για δύο-τρία χρόνια κατόπιν για να αντισταθμιστεί κατά κάποιον τρόπο όλο αυτό το φαινόμενο πρέπει να υπάρχει έλεγχος των εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών. Και τρίτον, αυτό σημαίνει ότι φτάνουμε σε περισσότερο πολιτική ενοποίηση. Και ε, περί αυτού πρόκειται, φτάνουμε στο διατάφτα. Το θέμα είναι ποιος έχει τις αρμοδιότητες, ποιος μπορεί να δώσει αυτή την εντολή τα κρατημέλη, τα εθνικά κοινοβούλια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εδώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει σημαντική αλλά περιορισμένη εντολή. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι αρμόδια για την σταθερότητα των τιμών και των χρηματοψηφιστικών αγορών. Καλή και σωστή η αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα, αλλά περιορισμένη. Αν όλοι οι άλλοι άμεσα εμπλεκόμενοι δεν διαδραματίζουν το ρόλο που του ανήκει, είναι πολύ δύσκολο για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να επιτύχει το στόχο, να συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου. Ευχαριστώ. Έχω μια πολύ σύντομη ερώτηση γιατί έχουμε εξαντλήσει κάπως το χρόνο μας. Σε ορισμένες από τις απαντήσεις σας αναφερθήκατε στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και όσο γίνεται αυτό να είναι σε επίπεδο 27 κρατών είπατε. Και ενδεχομένω ορισμένα ζητήματα παραδεχτήκατε ότι θα πρέπει να γίνουν σε επίπεδο 17 όπου το διακύβευμα είναι η σταθερότητα του ευρώ με περίεργη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω σε επίπεδο 17 τι θα μπορούσε να γίνει. Εντάξει, το θέμα για την επίλυση της κρίσης και τα τραπεζικά, αλλά γενικότερα στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες τι θα μπορούσε να υλοποιείται σε επίπεδο 17. Εννοώ ότι ο μόνος λόγος να γίνονται σήμερα ορισμένα στο επίπεδο των τώρα 17 κρατών είναι η προστασία του κοινού γενιαίου νομίσματος και η σταθερότητα των τιμών. Εγώ θα ε, καταβάλω κάθε προσπάθεια να κάνω ε, ό,τι μπορώ σε επίπεδο 27, αλλά γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι οι μεγάλα κέντρα βρίσκονται εκτός ευρωζώνης για το προσεχές μέλλον και το προβλέψιμο. Υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο γενικά παραγνωρίζεται όταν γίνεται λόγος για τη διαδικασία άρσης των ανισορροπιών. Κάτι που ρώτησε ο κύριος Κλούτε προηγουμένως. Η διαδικασία άρσης των ανισορροπιών έχει να κάνει με την καρδιά της οικονομικής πολιτικής. Δεν είναι απλώς δημοσιονομική πολιτική. Έχετε δίκιο γιατί ε, ήταν σφάλμα και αποτυχία του Συμφώνου Σταθερότητας να ασχοληθεί με τη δημοσιονομική πολιτική. Αν όμως το φέρουμε έτσι στα άκρα και συντονιστεί η οικονομική πολιτική στη συγκεκριμένη κατάσταση στην Ευρωζώνη με αυτές τις ανισορροπίες, κάποια στιγμή φτάνει κανείς στα όρια ε, και συγκρούεται με την εσωτερική αγορά. Δηλαδή, όταν τώρα πήξουμε στα άκρα και πούμε χρειάζεται συντονισμό, οικονομική μας πολιτική, ε, σε σχέση και με τις ανισορροπίες που έχετε δίκιο, δεν έχετε μόνο τη δημοσιονομική πολιτική των μελών της Ευρωζώνης. Και στην ακραία περίπτωση, και το γνωρίζουν οι συνάδελφοι στο Λονδίνο, μπαίνουμε στα χωράφια της ε, ε, ενιαίας αγοράς. Και αυτό είναι μια συνέπεια ε, την οποία αθέλητα έχει μια οικονομική πολιτική στο συντονισμό της. Σε ό,τι αφορά την οικονομική σταθερότητα, θέλω οι κανόνες όσο γίνεται να είναι για τους 27, για να εκμεταλλευόμαστε πλήρως τα ωφέλη της ε, κοινή αγοράς. Αλλά ταυτόχρονα χρειαζόμαστε κανόνες, ρυθμίσεις και εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο 27 κρατών. Αυτό γίνεται καλύτερα για όλες τις διασυνοριακές δραστηριότητες. Είναι καλύτερα σε επίπεδο 27 ή 16 ε, συν η εγχώρια αγορά του καθενός. Δηλαδή χρειάζεται σαφέστατα ε, ε, σταδιακή και βαθμιαία συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και με όλους τους μηχανισμούς. Οι ε, ε, χρηματαγορές χρειάζονται ρύθμιση σε επίπεδο 27 ή μήπως για την προστασία του ενιαίου νομίσματος έχει νόημα να γίνει αυτό σε επίπεδο 17. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι μια κλειστή λέσχη. Όποιο ε, θέλει και μπορεί, είναι και οι δύο όροι, να ενταχθεί στην Ευρωζώνη, ε, εντάσσεται. Ακόμα δεν κατάλαβα τι εννοείται, λέει η Πρόεδρος. Ε, ε δεν ξέρω, ίσως το δείξει ο χρόνος. Ε, ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλώς στις απαντήσεις σας σταθήκατε. Τώρα θα πρέπει να σας πούμε να εξέλθετε τις εθνούσεις και σε όλους τους άλλους που δεν δικαιούνται να είναι στην κεκλεισμένα των θυρών για να αποφασίσουμε για τη μοίρα σας. Ευχαριστώ πολύ.